ανάπτυξη δημιουργία θέσεων εργασία είναι κάτι που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Σα ευχαριστώ. Ωραία και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε και εσάς ε, για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Άρα λίγη συζήτηση επί αυτού του θέματος και Στη συνέχεια έχουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε σχέση με την εξέβρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Καταρχήν θα λάβει το λόγο ο κύριος Νικολάη Βάμεν, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κύριοι Επίτροποι, εξ ονόματος της ε, Δανέζικης Προεδρίας θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα, δηλαδή την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής. Πιστεύω ότι η η συνεργασία φορολογικών θεμάτων είναι προτεραιότητα για εμάς, ιδιαίτερα στα πλαίσια του παρόντος οικονομικού κλίματος, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να προωθήσουν την ε, δημοσιονομική εξυγίανση. Το Συμβούλιο έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει αυτή τη, αυτό το πρόβλημα αυτά τα χρόνια. Το 2006 και 2007 έφτασε σε συμπεράσματα για μια στρατηγική καταπολέμηση της φορολογικής απάτης σε κοινοτικό επίπεδο και έκτοτε το Συμβούλιο έχει εγκρίνει μία σειρά πράξεων όπως ε, την ε, μεγαλύτερη συνεργασία των κρατών μελών σε σχέση με την οδηγία VHE έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τις φοροαπαλλαγές και την καταβολή του ΦΠΑ στις εξαγωγές. Έχουμε λοιπόν προωθήσει και διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολόγησης έτσι ώστε να υπάρχει αμοιβαία αρρωγή για την αποτίμηση των διαφόρων φόρων και φορολογικών βάσεων μεταξύ κρατών μελών και ανταλλαγή πληροφοριών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, το 2003 ε, ελήφθη υπόψη μία οδηγία σε σχέση με τις αποταμιεύσεις και επίσης αμοιβαία αγωγή σε σχέση με αξιώσει, σε σχέση με, τις, ε, με τα φορολογικά μέτρα, τέλη και δασμούς που έχουν καταβληθεί. Νομίζω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δείχνουν την δέσμευση του Συμβουλίου να καταπολεμήσει την φοροδιαφύγη και την ε, καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Πέρσι το Μάρτιο τονίσαμε τη σημασία της ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης και γι' αυτό Ζητήθηκε από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να βρουν τρόπους για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, έτσι ώστε φέτος τον Ιούνιο να αποτιμήσουμε την κατάσταση. Η Προεδρία της Δανίας προσδίδει μεγάλη σημασία σε αυτό το ζήτημα και προωθείται αυτή η εργαστία. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε θέση τον Ιούνιο να ανταποκριθούμε στο αίτημα του Συμβουλίου. Βεβαίως σε αυτό το στάδιο δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει αυτή η έκθεση. Μπορώ όμως να σας μιλήσω για την εργασία του Συμβουλίου, για την τρέχουσα εργασία. Καταρχήν η Ιδανική Προεδρία ε, ο, προωθεί ε, μία οδηγία που θα στηθεί από το ΕΚΟΦΗΝ το Μάιο-Ιουνίο σε σχέση με τις αποταμιεύσεις. Επίσης θα οριστεί εντολή έτσι ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης για μία νέα γενεά φοροαπαλλαγών ή φοροαποταμιεύσεων. Και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη την φορολογική βάση και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για να μπορέσουμε να προβούμε σε διασυνοριακές αποταμιεύσεις. Πιστεύουμε ότι θα επιτελεστεί πρόοδος σε αυτό το δύσκολο θέμα, το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης σε σχέση με την οδηγία για την διοικητική συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών θα εγκριθεί κατά το επόμενο ΕΚΟΦΗΝ έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη. Σε σχέση με τον ΦΠΑ θα ναι. υπάρξει ειδική ανακοίνωση της Επιτροπής και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα στο τέλος της ε, Προεδρίας ε, της Δανίας. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας για τον συντονισμό των φορολογικών πολιτικών και η ομάδα του Συμβουλίου ε, οδηγείται, μάλλον λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα για να προωθήσει μία νέα βάση φορολόγησης των επιχειρήσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα συνεργαστούμε μαζί σας και με την Επιτροπή έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστεί και ο Πρόεδρος. Και τώρα έχει το λόγο ο Επίτροπος Σεμέτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, στη δύσκολη αυτή εποχή που ζούμε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι φόροι θα συλλέγονται δίκαια και σωστά. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους πολίτες να δεχτούν πρόσθετα βάρη φορολόγησης εάν δεν κάνουμε πρώτα ό,τι μπορούμε για να περικόψουμε δαπάνες και πρακτικές που τους μειώνουν το εισόδημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε βελτίωση επ' αυτού. Το περασμένο Δεκέμβριο είχαμε πει ότι ήδη επεξεργαζόμαστε μια στρατηγική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής το αίτημα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και το σημερινό σας αίτημα μας δίνουν μια περιττέρω όθηση. Γι' αυτό θέλω να ακούσω σήμερα τις απόψεις σας. Για να πλαισιώσουμε καλύτερα μια τέτοια ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τρία θέματα. Πρώτον, τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση των υπαρχών των εργαλείων. Παραδείγματο χάρη το Ευρωφίσκ θα μπορούσε να δώσει πραγματικές πληροφορίες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και να κάνει καλύτερες αξιολογήσεις. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Eurofisk και το πρόγραμμα Fiscalith. Στην άμεση φορολόγηση πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους μηχανισμούς που προτείνονται. Και αυτό με βγει στο δεύτερο θέμα. Η πρόοδος στο Συμβούλιο για τις εκκρεμούσες προτάσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής ναι. είναι, η πρόοδος αυτή είναι πολύ αργή. Πρέπει να βρουν οι υπουργοί έναν τρόπο να βγουν από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται για πάρα πολύ καιρό ως προς την αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας την για την αποταμίευση. Πόσο μάλλον που οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις το δείχνουν ακόμη περισσότερο. Δεν υπάρχει σχεδόν πια το τραπεζικό απόρριτο. Είναι καιρό η Ένωση να δημιουργήσει δικούς της μηχανισμούς. Και ο πρώτος τέτοιος θα ήταν το Συμβούλιο να ζητήσει από την Κομισιόν να διαπραγματευτεί με τους εταίρους μας, ιδιαίτερα με την Ελβετία. Έπειτα. Πρέπει να υπάρξουν καινούργιε ιδέε. Τι δηλαδή. Παραδείγματο χάρη μια κοινή προσέγγιση για τις έρευνες όχι μόνο διαμεθοριακός αλλά και μεταξύ διαφόρων οργάνων όπως τα τελωνία και τις εφορίες. Ένας νέος μηχανισμός που να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αντιδράσουν εγκαίρως όταν διαπιστώνονται απάτες εις βάρος της ίσπραξης του ΦΠΑ. Επίσης θα ήθελα να υπάρξει μεγαλύτερη καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Πρέπει να βρούμε τρόπο πολιτική θέληση για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε, θα, θα μπορούμε να αμυνθούμε έναντι όσων δεν εφαρμόζουν τους κανόνες. Αυτή τη στιγμή γίνεται η σχετική διαβούλευση και θα κάνω ό,τι μπορώ για να καταπολεμηθούν οι πρακτικές που εμποδίζουν την συλλογή του φόρου. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε ότι χρειάζονται βελτιώσεις όχι μόνο στη φορολογική νομοθεσία ως Επίτροπος Αρμόδιος για την καταπολέμηση των απατών, τον περασμένο Ιούνιο καταστρώσαμε την αντιαπατική στρατηγική της Κομισιόν όπου είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τη χρήση και δαπάνηση των ε, νοσιακών πόρων και ταμείων. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο δεν θα δέχονται πια επιχορηγήσεις. Ο συνάδελφός μου Μισελ Μπαρνιέ επίσης είναι πολύ δραστήριος έχοντας κάνει πρόσφατες προτάσεις για καλύτερη πληροφόρηση της δραστηριότητας των εταιριών. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αντιδρούμε στεναρά για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής και προσδοκώ σε μια επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα έχουν το λόγο οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων για το ΕΛΚ Ζάλβα Το... Στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίστηκε η ανάγκη να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα καταπολεμώντας κυρίως τη φοροδιαφυγή. Και η Ισπανία εκπώνησε ένα σχετικό νόμο. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου αποτελούν προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της Ισπανίας και της υπόλοιπης Ευρώπης κατά συνέπεια. Θα έχουμε νομική ασφάλεια. Θα καταφέρουμε να μειώσουμε την παραοικονομία και να καταπολεμήσουμε όσους φοροδιαφεύγουν. Θα έχουμε κατά συνέπεια μια Ευρώπη πιο δίκαια. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις συστάσεις του ΩΣΑ για να μειώσουμε τις διαφορές μεταξύ όσων πληρούν τα, τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και όσων δεν τις πληρούν. Εμείς θα υπερψηφίσουμε τα οποία θέλουν διαφάνεια και συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επιτρέψουν να μειώσουμε το έλλειμμα και δεν θα προδικάσουν τις αναπτυξιακές συνθήκες. Θα δημιουργήσουν ένα σύστημα πιο δίκαιο το οποίο θα βελτιώσει γενικά τις ευκαιρίες και θα βοηθήσει στην ανόρθωση των δημοσιονομικών. Θα μειώσει το έλλειμμα, όπως σας είπα, και θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη. Και επειδή μιλάμε για ανάπτυξη, δεν θα ήθελα να μην αναφέρω ότι θα πρέπει να παλέψουμε για την διεθνοποίηση της οικονομίας μας και των επιχειρήσεών μας, όπως το δήλωσε και το Συμβούλιο πολλές φορές. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να εγγυθούμε την νομική ασφάλεια των επενδύσεών μας. Και δεν θέλω να προδικάσω τη συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να απαντήσετε σε μια ερώτηση με μπλε κάρτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σάλμπα, αναφερθήκατε πολλές φορές στα κυβερνητικά σχέδια στην Ισπανία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αναφέρεστε ίσως το σχέδιο της Ισπανικής κυβέρνησης για την γενική αμνηστία φορολογική αμνηστία για τους ε, φοροδιαφεύγοντες. Λοιπόν, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτόν τον νόμο σας παρακαλώ. Κυρία Μουνής, καταρχήν να σας πω ότι καμία φορολογική αμνηστία δεν ενεκρίθη από την Ισπανική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο Ισπανικό Σύνταγμα. Η Ισπανική κυβέρνηση μια ρύθμιση πρότεινε όπως κάνανε και άλλες χώρες, Βέλγιο ή Ισπανία για παράδειγμα. Οι άλλες κυβερνήσεις ισπανικές ε, του ιδίου πολιτικού σας χρώματος, δηλαδή σοσιαλιστικές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους ε, σοσιαλιστές. Ε, έχει τώρα το λόγο η κυρία Φεραίρα. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ βαριά για τους Ευρωπαίους πολίτες όλη αυτή η ιστορία ανόρθωσης των προϋπολογισμών Πολλοί υποφέρουν από αυτά τα μέτρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, καταναλωτές, όλα αυτά πέφτουν στην πλάτη τους και παράλληλα έχουμε μια τεράστια φοροδιαπηγή. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να ξέρω ποιο είναι το ποσό που υπολογίζεται στις 27 χώρες. Ένα τρισεκατομμύριο παραπάνω από όσο ξοδεύουμε ένα δις δηλαδή παραπάνω από όσο ξοδεύουμε για την υγεία. Μάλιστα. Αν εμείς ε, πιάναμε το 1 πέμπτο αυτού του ποσού, θα περνάγαμε σε ένα 3,5% επενδύσεων. Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό. Το ψήφισμα το οποίο θα εγκρίνουμε θέλει να στείλει αυτό το μήνυμα της απέτηση δηλαδή, ώστε Συμβούλιο και Κομισιόν να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες φορολογικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις όμορες χώρες, πιο συγκεκριμένα με την Ελβετία, διαπραγματευμένες όμως από την Κομισιόν, όχι χώρα με αναχώρα διμερός. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τους ε, κανόνες υπολογισμού. Θα πρέπει να, να αυξήσουμε τη διαφάνεια. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι... το πρόβλημα των φορολογικών παραδείσων για να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή. Στα πλαίσια των G20 θα πρέπει να ξεκινήσουμε έναν κοινό αγώνα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αυτό είναι έντιμο για τους πολίτες μας. Τελευταία μου λέξη λοιπόν. Ας παλέψουμε ούτως ώστε Συμβούλιο και Κομισιόν να προχωρήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Σας Παίρνω το λόγο για να εκφράσω τη συμφωνία μου με αυτό το ψήφισμα και τα μέτρα. Η καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής αποτελεί απόδειξη θεσμικής αποτελεσματικότητας και ηθικής υποχρέωσης. Βελτιώνει τα δημοσιονομικά και χτυπάει τους απατεώνες. Ενισχύει την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη βάσεις της συμβίωσής μας. Σύμφωνο ότι η φορολογική εναρμόνιση, ο συντονισμός των ευρωπαϊκών θεσμών και των Ευρωπαϊκών Υπουργείων Οικονομικών είναι σημαντικότατη. Η περιφέρειά μου, η οποία είναι φορολογικά αυτόνομη, επλήγει διότι ε, χρησιμοποίησε φορολογικά μέτρα που χρησιμοποιούν άλλες χώρες οι οποίες όμως ποτέ δεν επιπλήχθησαν γι' αυτό. Πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία για να καταπολεμήσουμε και τον αθέμητο ε, ανταγωνισμό και τη φοροδιαφυγή με συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης θα ήθελα να συμμεριστούμε τις καλές πρακτικές για να συμμεριστούμε και οι πολίτες αυτήν την κοινή αξία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την διαφθορά, άλλη πληγή στη δημόσια διοίκηση. Ευχαριστώ για τους ε, πράσινους, ο κύριος Γκίγκολτ. Ναι, Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και της οικονομίας στην Ευρώπη δεν αφήνει περιθώρια για φορολογικά παραμύθια. Οι φορολογικές προτάσεις δεν προχωρούν. Γιατί? Γιατί κάποιες χώρες είναι κατά της περαιτέρω συνεργασίας. Εποφελούνται από την κατάσταση είναι φορολογικές οάσεις και αναφέρεται στις συνθήκες πως τα φορολογικά απαιτούν ομοφωνία. Οπότε κομισιόν στο παρελθόν ε, οδηγείται σε ναυάγια με τις προτάσεις της. Τίποτα δεν προχωράει. Και πλέον έμαθω μαθημάτης και δεν προτείνει τίποτα το φιλόδοξο. Ξέρω κύριε Σεμέτα πως είναι δύσκολη η δουλειά σας. Αλλάξτε όμως τη στρατηγική σας. Προτείνετε σκληρά μέτρα και ε, φροντίστε να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία για να ξεπεράσετε το μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο. Europos ekonomikos ir ūkio nuosmukio kontekste mokesčių surinkimas ir jų politikos klausimai įgauna ypatingą svarbą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 Και έχουμε άλλες πολυεθνικές επιχειρήσεις ευρωπαϊκές, οι οποίες, μάλλον και η Coca-Cola είναι Ολλανδική και η IKEA είναι Ολλανδική στην Ολλανδία, όλα αυτά με διοικητικά γραφεία στην Ολλανδία και με βάσεις παντού στο εξωτερικό. Και υπάρχει συμφωνία με το Ολλανδικό κράτος και πληρώνουν όσο το δυνατόν λιγότερο φόρους πληρώνουν ελάχιστο φόρο στην Ολλανδία και τα κέρδη τα στέλνουν στους ε, φορολογικούς παραδείσους. Είναι πραγματικά απαγοητευτικό να βλέπει κανείς τέτοιου είδους ε, ε, με μεγάλο επιχειρήσεις, πολυεθνικές επιχειρήσεις να φοροδιαφεύγουν όταν ο κόσμος στην Ευρώπη σφίγγει το ζωνάρι του. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επέμβει. Στο ψήφισμα ζητούμε εμεί διαφάνεια. Οι ετήσιοι λογαριασμοί των πολυεθνικών να είναι ακριβέστερη χώρα προ χώρα να μπορούμε να ελέγχουμε τον κύκλο εργασιών και να γίνεται δίκαια φορολόγηση. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μία ακτινογραφία της κατάστασης, μία χαρτογράφηση και να καταλήξουμε να έχουμε μια δίκαιη φορολόγηση. Ελπίζω λοιπόν να το υποστηρίξει η Κομισιόν. Κύριε Ποδηματά. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, πήραμε την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είναι και πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα και των εθνικών και των ευρωπαϊκών στρατηγικών εξόδου από την κρίση γιατί η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή καθιστούν κοινωνικά άδικο τον επιμερισμό του κόστους και υπονομεύουν για λόγου οικονομικούς και κοινωνικούς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. είναι παραλογισμός να προχωράμε την εμβάθυνση μόνο στη δημοσιονομική πολιτική χωρίς να κάνουμε αντίστοιχα βήματα σύγκλησης και συντονισμού της φορολογικής πολιτικής με αποτέλεσμα να ενισχύεται ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ μας και να επιδεινώνονται τα δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. και δεν είναι μόνο ο μεταξύ μας φορολογικός ανταγωνισμός είναι και η φυγή κεφαλαίων προς το εξωτερικό προς την ελβετία αλλά και προς άλλες χώρες μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης που ακόμα διατηρούν το τραπεζικό απόρριτο. προφανές είναι ότι υπάρχουν εθνικές ευθύνες για τη φοροδιαφυγή το ίδιο ισχύει και για τη δημοσιονομική κρίση αυτό όμως δεν εμπόδισε το συμβούλιο και την επιτροπή να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες και πολιτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 15 Μαΐου θα πρέπει να αγωνιστούμε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή εντολή προς την Κομισιόν. Αυτό είναι καλό από την πλευρά του Συμβουλίου. Μπορούμε να καταμετρήσουμε στη συνέχεια σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ελβετία και άλλες χώρες έχει καταφέρει να διαπραγματευτεί κάποιες λύσεις. Αλλά θα είναι πολύ σωστό να πούμε και στους συναδέλφους ότι πρέπει να βασιστούμε στην ενισχυμένη συνεργασία. Αυτή τη στιγμή περιμένει κοινή γνώμη από εμά να υπάρξει μια απάντηση. Ρωτήστε τη γερμανική κυβέρνηση, ρωτήστε την γαλλική κυβέρνηση, γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα. Γιατί παρά τα λόγια τους δεν έχουν προχωρήσει σε πρωτοβουλίες. Και απαντήστε επίσης και στο ερώτημα γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πολύ πιο επιτυχημένοι στις διμερείς συμφωνίες που έχει κάνει, απλώς γιατί μπορεί να ασκήσει πίεση παραδείγματο χάρη στην Ελβετία, περισσότερη πίεση από ό,τι μπόρεσε να ασκήσει η γερμανική κυβέρνηση. Σκεφτείτε λοιπόν και πάλι τα συμφέροντα των πολιτών, γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνει κάτι διαφορετικό και καταφέρνει σε πρακτικό επίπεδο να επιτύχει του στόχους της. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Η φοροδιαφυγή προκαλεί τεράστιες οικονομικές απώλειες. Επηρεάζει τη λειτουργία των θεσμών του κράτους και θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Η Ρουμανία έχει ένα μεγάλο ποσοστό του, ελ, του, το οποίο μπορεί να φτάνει και το 40% το οποίο διαφέρει με τον τρόπο αυτό. Είναι απαραίτητο να, να αγωνιστούμε εναντίον τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή και υπάρχει και μια πρόταση για το Συμβούλιο των Υπουργών Συνεδρία σε σχέση με το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και ερωτήματα για τη παραμονή της Ολλανδίας στην χώρα, στον χώρο του Σέγγεν. Και αυτό έχει να κάνει με, τις, ε, με τη λαθρεμπορία που λαμβάνει η χώρα. Και υπήρξαν προϊόντα τα οποία μπήκανε στο λιμάνι του Ρότερνταμ χωρίς κανένα έλεγχο. Και την ε, προηγούμενη εβδομάδα ανακαλύφθηκαν αντίστοιχες απάτες από τις Ιρλανδικές αρχές. Ο κύριος Χρυσαγκέλτος έθεσε ένα, μια μπλε κάρτα. Θέλετε να θέσετε ένα ερώτημα στην κυρία Μπασέσκου. επισημάνω και να ρωτήσω τον κύριο επίτροπο η ελλάδα όπω ξέρουμε αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. από την άλλη μεριά όμω ξέρουμε ότι υπάρχουν σε ελβετικέ τράπεζε Συγγνώμη, ε, δεν είναι αυτή η διαδικασία της μπλε κάρτας. Η μπλε κάρτα μπορεί να σας επιτρέψει να θέσετε ένα ερώτημα σε κάποιον άλλο βουλευτή, ο οποίος μόλις είχε πάρει το λόγο. Μόνον έτσι, δεν είναι αυτή η διαδικασία λοιπόν. Ακολουθούμε τη διαδικασία catch the eye, όπως λέμε στα αγγλικά. Και τώρα δίνω το λόγο, κύριο Ζάνκα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι σε σχέση με τη χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη είναι πολλά τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν αυξήσει τη φορολογία τους. Αλλά αυτός είναι ο λαφασμένο τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τροχοπεδείται η ανάπτυξη στον οικονομικό χώρο και σίγουρα δεν δημιουργούνται νέε θέσει απασχόλησης. Μια πολύ βελτιότερη στρατηγική θα ήταν να βελτιώσουμε την ίσπραξη των φόρων και η αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε μικρότερο οικονομικό αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία και έτσι μπορούμε να αυξήσουμε και την ανταγωνιστικότητα των χωρών μας. Εγώ έχω ακούσει πολλά στη σημερινή συζήτηση και ανησυχώ ως εκ τούτου. Βλέπω ότι δεν υπάρχει μια αποφασιστική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τη στιγμή όμως που η Ευρώπη βρίσκεται σε μια οικονομική στενοπό, χρειαζόμαστε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση. Ο κύριος Καλπέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα επίκαιρο θέμα πράγματι. Η απόκρυψη, και... απόκρυψη φόρων και φοροδιαφυγή είναι τεράστιες οι επιπτώσεις. Σε έχει πλήξει ιδιαίτερα η οικονομική κρίση και αντί να αποδιόμεθα σε οράματα και όνειρα, θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην ίσπραξη των φόρων και πιο πραγματιστικοί. Αν δεν το πράξουμε αυτό, τότε οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αποσύρουν την ε, υποστήριξή τους και την εμπιστοσύνη τους προς εμάς. Γι' αυτό αυτή η πρωτοβουλία είναι αξιοσημείωτη. Το να υπάρξει μια καλύτερη διαδικασία ελέγχου των διμερών συμφωνιών θα είναι ιδιαίτερα επωφελές, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση της φοροδιαφύγης. Έτσι, τα λεγόμενα υβριδικά μέσα, τα οποία έχουν ε, παρουσιαστεί. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Ο κύριος Πόσελτ. Η αντιμετώπιση της ε, φοροδιαφυγής και φοροαπάτης έχει μεγάλη σημασία γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία ελείπουν από τον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν σε μέτρα αναπτυξιακά στις χώρες αυτές και επομένως θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αντιμετώπιση της κρίσης. Το να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στα κράτη-μέλη και μια καλύτερη <clears throat> συνεργασία μέσα στα πλαίσια του άρθρου 65 είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Παπα-Νικολά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 1% του ΑΕΠ της, Ευρώπης κοστολογείται η φοροδιαφυγή και η διαφθορά περίπου δηλαδή 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, με πρόσφατη αξιολόγηση επίσης τα, 3 πέμπτα, τα 2 τρίτα με των κρατών μελών ε, της Ευρώπης απέτυχαν σε πρόσφατη αξιολόγηση να πάρουν βαθμό πάνω από 5 στα 10 για τα θέματα της διαφθοράς. Το λέω αυτό για να πω και για τη φοροδιαφυγή ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο για κάποια κράτη μέλη όπως συχνά αναφέρουν κάποιοι συνάδελφοι είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό και ω τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. πέραν των όσων υπόθηκαν από του συναδέλφου θα ήθελα να προσθέσω μια ακόμη παράμετρο πολύ σημαντικά κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι αφιερωμένα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. ένα δισεκατομμύριο περίπου είναι αφιερωμένο για την ελλάδα μέχρι το 2013... σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την αναμόρφωση τη δημόσια διοίκηση. αυτού του πόρου του αξιοποιούμε στοχευμένα στην καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή; αυτή είναι η ερώτησή μου προ την κομισιόν και το συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σεμέτα για να κλείσει τη συζήτηση. Uh, Αγαπητά μέλη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι η συζήτηση ήταν επικοδομητική και επίκαιρη. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τις απόψεις που εκτέθησαν και πράγματι θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά τις απάτες γύρω από τη φορολογία και τη φοροδιαφυγή. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υπογράμμισαν τη σημασία της δράσης στο συγκεκριμένο τομέα. Η πρόκληση είναι αυτή η πολιτική βούληση να γίνει πραγματικότητα. Τα αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα αποτούν, απαιτούν πολλά πράγματα. Σωστό σχεδιασμό, αποτελεσματικούς ελέγχους. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επεξεργαστούν και να αντιμετωπίσουμε φυσικά και τα θέματα της φυγής των κεφαλαίων εκτός χώρας. Αυτά θα εξεταστούν και στα πλαίσια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και έτσι στα πλαίσια του θέματος της οικονομικής διακυβέρνησης θα εμείνουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή γύρω από το θέμα της καταπολέμησης της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Δύο βασικές προτεραιότητες. Πρώτον, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο τον μήνα Ιούλιο θα είναι μια σωστή και ρεαλιστική βάση για περαιτέρω εξελίξεις. Έχει μεγάλη σημασία να κινητοποιήσουμε τους Υπουργούς Οικονομικών να αντιμετωπίσουν τα θέματα γύρω από τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Δεύτερον, θα εκθέσουμε τους επόμενους μήνες και τις απόψεις μας για την πρωτοβουλία την οποία θέλουμε να πάρουμε σε σχέση με τις λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους. Σήμερα μου δώσατε ένα εξαντλητικό θα έλεγα κατάλογο ανησυχιών κυρίως και ιδεών. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε και στην συμφωνία με την Ελβετία. Και εγώ εδώ προσβλέπω στις προσπάθειες της Προεδρίας της Δανίας έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ανοίξει ο δρόμος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί με την Ελβετική Ομοσπονδία και να δώσει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να συλλέξουν τους φόρους για τα χρήματα που έχουν διαφύγει. Κάποιοι από εσά <clears throat> αναφερθήκατε και στα θέματα του επιθετικού φορολογικού ε, λεγόμενου προγραμματισμού και θα κάνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου <clears throat> για την σωστή χρήση των ορθών πρακτικών και την κυκλοφορία των ορθών πρακτικών. Έχουμε πάρει ήδη πρωτοβουλίες στα πλαίσια του φόρουμ που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητάμε από τα κράτη-μέλη να μοιραστούν τις πρακτικές τους, τις ορθές πρακτικές τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα κράτη-μέλη. Ο κ. Μπούλμα έθεσε το θέμα της ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της καταπολέμησης της φορολο... και φοροδιαφυγής. Δεν είμαστε χειρότεροι από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θέλουμε όμως να συνεργαστούμε περαιτέρω με τις Ηνωμένε Πολιτείε και να προωθήσουμε στοιχεία και πληροφορίες για καλύτερη ενημέρωση αμοιβαία και πληροφόρηση αμοιβαία και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά όχι μόνο στα πλαίσια της σχέσης μας με την Ελβετία αλλά και με άλλες τρίτες χώρες για τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εμπλεκομένων σε σχέση με τα θέματα τα φορολογικά. Εδώ η υποστήριξη του Κοινοβουλίου έχει μεγάλη σημασία αν θέλουμε να προχωρήσουμε και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο στήριξης των νομοθετικών πρωτοβουλειών. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κύριε Υπουργοί, με μεγάλη χαρά πήρα μέρο και ε, νομίζω ότι συνεισέφερα στη σημερινή συζήτηση. Από πλευρά μου, εγώ εξετίμησα δεόντως την συνεισφορά σα και αναμένω περαιτέρω δυνατότητε και ευκαιρίες συζήτηση αυτού του τόσο σημαντικού θέματος. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Βάνεν από το Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, επίτροπε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν τη συζήτηση η οποία αποδεικνύει ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής βρίσκονται στην καρδιά των τριών θεσμικών οργάνων. Εμείς επιμένουμε ιδιαίτερα σε αυτό το ζήτημα. Εμείς στις τοποθετήσεις μας σήμερα υπογραμμίσαμε την σημασία που δίνουμε σε αυτό το θέμα. Θέλω να δράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Σεμέτα που έκανε μια ανασκόπηση των ε, επεμβάσεων της ε, Κομισιόν στον τομέα και εμείς ως ε, Δανική Προεδρία προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με τον Επίτροπο και την Επιτροπή. Στην αρχή της τοποθέτησής μου είπα ότι υπάρχει μία ολόκληρη πανοπλία ε, προτάσεων που συζητιούνται σήμερα στο Συμβούλιο και τα αποτελέσματά τους θα γίνουν ορατά στο εγγύς μέλλον. Το θέμα της Ελβετίας ε, θύχθηκε. Η Δανέζικη Προεδρία επιμένει ούτω ώστε να δοθεί σύντομα εντολή για να διαπραγματευτούμε μία συμφωνία με την Ελβετία. Σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και με την Κομισιόν η Προεδρία θα κοιτάξει να επιταχύνει τα πράγματα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προοδεύσουμε σε αυτά τα θέματα, κυρίως όσον αφορά στην φορολόγηση των εισοδημάτων. Ε, ελπίζω ότι θα πετύχουμε πολλά και γρήγορα. Θα θέλαμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ακολουθήσει τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έθεσε αυτό το σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η Δανική Προεδρία μαζί με το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να προοδεύσουμε στα θέματα αυτά και η φοροδιαφυγή και η καταπολέμησή της να είναι στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ημερήσιας Διάταξης, ούτως ώστε όλοι να συνεισφέρουμε στην κοινοτική ευημερία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Έχω ένα ψήφισμα ενώπιον μου το οποίο έχει υποβληθεί. Κλείνουμε τη συζήτηση και η ψήφιση αυτού του ψηφίσματος θα είναι την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη δήλωση